Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, όλες τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί θα διαβιβαστούν στους αποδέκτες σας. Σας παρακαλώ. Ναι, αν θέλετε διαδικαστικά να παρέμβετε, ευχαρίστω. Κύριε Πρόεδρε, για να σας πω την αλήθεια, εγώ εκπλήσωμαι με τον τρόπο με τον οποίο έχετε συμπεριφερθείτε σήμερα. Φυσιολογικά είσαστε πάντα πολύ σωστός σε ό,τι αφορά το χρόνο αγόρευση Αλλά η συμπεριφορά σας σήμερα είναι ακατανόητη για μένα. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και είναι παράξενο το ότι τέθηκε σε τέτοια χρονική στιγμή στο απόγευμα της Πέμπτης και τώρα περικόπτεται τη συζήτηση. Μετά από 18 λεπτά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί. Κυρία Γιασοβλέκα. Η συνέλευση των Πρόεδρων είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά. Κύριε Καμπούτο, θα σα δώσω το λόγο αμέσω. Είναι η συνέλευση των Πρόεδρων αρμόδια να καθορίσει την ημερήσια διάταξη. Το ότι έχουμε τελειώσει λίγο νωρίτερα οφείλεται στο, ότι, στο γεγονός ότι στην προηγούμενη συζήτηση δεν υπήρξε καθόλου δια, δι, χρήση του χρόνου catch the eye. Εγώ θα ήθελα ο κύριος Καπούτο μπορεί και αυτό να θέλει να, να διαμαρτυρηθεί Λοιπόν, κύριε Καπούτο, αν θέλετε και το λόγο, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, εγώ θέλω απλά να καταλάβω το κριτήριο. Εσεί δώσατε το λόγο σε 8 ανθρώπους ανάμεσα στο Άλντε και το ΕΛΚ. Μόνο εγώ σας ζήτησα το λόγο από τους σοσιαλιστές και δεν μου δώσατε και το λόγο και μάλιστα δικαιολογηθήκατε λέγοντας ότι δεν θα δίνατε το λόγο σε όσους προηγουμένως το είχαν λάβει. Εγώ ε, δεν το είχα λάβει το λόγο ενώ κάποιο άλλος ναι. Ε, είναι διάκριση αυτό και μάλιστα δικαιολόγητη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καπούτο. Θα ήθελα να σας πω σαφώς ότι κανείς δεν ζήτησε το λόγο από τη μεριά τη σοσιαλιστική ομάδα μετά ήρθατε εσεί. Στην αρχή δεν άφησα τον κύριο Τσαμπάσκι να λάβει το λόγο γιατί είχε μιλήσει ακόμα. Εγώ επομένως θέλησα να τηρήσω αυτή την αρχή ότι αυτοί που είχαν μιλήσει δεν θα λάμβαναν πάλι το λόγο. Δεν υπήρξε κάποιο άλλος λοιπόν ο οποίο από την ομάδα σα να ζητήσει. Είχαμε τρία μέλη από το ΕΛΚ και δύο από την άλλη, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δέκα που ζητήσαν το λόγο. Προσπάθησα να διατηρήσω μια ισορροπία και λίγη η συνεδρίαση.